Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε άμεσα. η είναι ε, ε, ε, κοινά η συνεδρίαση η οποία διεκόπη. Ο κύριος Στίβεν θέλει, ο κύριος Στίβενσον θέλει να μιλήσει νομίζω για την αντιπροσωπεία στο Ιράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τα νέα σήμερα το πρωί ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ε, απεκάλυψε μία συνωμοσύνη ε, των ε, Ιρανών να ε, δολοφονήσουν το Σαουδάραβα πρέσβη στη Washington ε, καθώς και ο αριθμός των ε, μελοθανάτων που φτάνει τα 13 άτομα στο Ιράν και σε άλλες πόλεις στην και σε άλλα σημεία είναι ένα θέμα που το η διάσκεψη των προέδρων θα πρέπει να εξετάσει και γι' αυτό αποφάσισε να στείλει σε δύο-τρεις εβδομάδες ε, ε, μία αποστολή διότι ε, το Ιράν αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατόν να κινείται έτσι και πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε την απόφαση που ελήφθη από τη διάσκεψη των προέδρων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βεβαίως η ε, παρατήρησή σας θα ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Σαλάτο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στο φως των ε, αυτών που μόλις ελέγχθησαν και επειδή εγώ είμαι μέλος αυτής της αντιπροσωπείας η οποία πρόκειται να πάει στην Τεχεράνη και μαζί με τους Ιταλούς συναδέλφους μας ε, αντιτιθέμεθα πλήρως στην ε, αποστολή αυτή στο Ιράν και θα ζητούσα από τη διάσκεψη των Προέδρων που έδωσε το πράσινο φως στην αποστολή αυτή ε, να αναθεωρήσει την απόφασή της διότι δεν θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Ιράν. Ευχαριστώ. Ε,